τη συζήτηση για ε, καταστάσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας και κράτους δικαίου. Θα μιλήσουμε για την ε, κατάσταση στις Μαλδίβες. Ξεκινούμε με τον συντάκτη, τον κύριο Κοράου. Κύριε Κοράου, έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το αρχιπέλαγος των Μαλδίβων δεν είναι το πολύ ωραίο ε, μέρος ε, με την καταγάλανη θάλασσα και τις ωραίες ακτές. Δυστυχώς πολλοί εργαζόμενοι από το Μπαγκλαντές και την Ινδία ε, την χάνουν εκμετάλλευσης και λαμβάνουν ψυχία έναντι αμοιβή. Επίσης υπάρχουν πολλοί πολιτικοί φυλακισμένοι υπάρχει κλίμα εκφοβισμού και τρομοκρατίας. Η κυβέρνηση παραβιάζει το διεθνές δίκαιο σε σχέση με, την, με τα βασανιστήρια. Επίσης παραβιάζονται τα δικαιώματα των γυναικών. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την επανεισαγωγή της θανατικής ποινής της Μαλδίβες. Θα θέλαμε να ε, διατρανώσουμε τη θέλησή μας κατά της θανατικής ποινής. Το δικαίωμα στη ζωή είναι το πολυτιμότερο αγαθό και θα πρέπει να μην δεχτούμε και τα βασανιστήρια και τον ψυχολογικό εκβιασμό. Λάμπερτ, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε λαμβάνω το λόγο ως ε, πρόεδρος αντιπροσωπής για τις σχέσεις με την Νότια Ασία, στην οποία εντάσσονται και οι Μαλδίβες. Συμφωνώ ότι η παρούσα κατάσταση στις Μαλδίβες ε, μας δημιουργεί τεράστιο προβληματισμό και ανησυχίες. Ακούσαμε την αναβίωση της θανατικής ποινή που από το 1950 δεν είχε χρησιμοποιηθεί στις Μαλδίβες και αυτό μας ε, ανησυχεί πάρα πολύ. Το Σύνταγμα έχει μόνο μία δεκαετή ζωή μέχρι στιγμής είχαμε μέχρι στιγμής μια δημοκρατική εξέλιξη, την οποία παρακολουθήσαμε εκ του σύνεγγυς, αλλά τώρα πια βλέπω μια υποχώρηση της δημοκρατίας, μια παλινδρόμηση και βασικά στοιχεία του δημοκρατικού συντάγματος, όπως η διάκριση των εξουσιών, παραβιάζεται. μεταξύ επίση ε, του Προέδρου και της δικαστικής εξουσίας. Ε, θέλουμε μια αμερόληπτη δικαστική εξουσία που όλοι είναι ίσοι έναντι του νόμου, ο νόμος εφαρμόζεται ισότιμα σε όλους και δεν ε, έχουμε νομοθετικές διατάξεις που προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, ε, συγκεκριμένων ιδιωτών και κυρίως του πρώην Προέδρου Νασίντ. Θα πρέπει επίσης να αναγνωριστεί από όλα τα πολιτικά κόμματα ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί η ποιότητα της δικαστικής εξουσίας. Και ισχυρά και ανεξάρτητα θεσμικά όργανα επίση είναι σημαντικά. Γιατί και η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει υποστεί επιθέσει, ε, τα μέσα μαζική ενημέρωση ε, φημώνονται και ο χώρο τη κοινωνία των πολιτών και τη δημοκρατική αντιπολίτευση όλο και συρρυκνώνεται. Όλα αυτά είναι πραγματικά εκτροπή προς τη λάθος κατεύθυνση για τις Μαλδίβες. Εξού και το ψήφισμά μας προκειμένου να ενθαρρύνουμε τις Μαλδίβες να ακολουθήσουν την πρόοδο προς τη σωστή κατεύθυνση. Κύριε Ντεπρέ, έχετε το λόγο για ένα λεπτό, ως εισηγητής. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Αντικαθιστώ τον κύριο Νάρτ που έχει καθυστερήσει. Υπάρχουν ε, ιδιαίτερες περιπτώσεις ε, ε, για παράδειγμα, όσοι έχουν επισκεφτεί τις ε, Μαλδίβες ε, έχουν την ιδέα ενός ιδηλιακού τοπίου του παραδείσου, αλλά βλέπουμε ότι είναι μια χώρα που το 2014 επανέφερε τη Σαερία, τον Ισλαμικό νόμο και με εφαρμόζεται θανατική ποινή ακόμη και σε παιδιά από 7 χρονών. Μάλιστα, ένας ε, ανήλικος που έχει καταδικαστεί σε θάνατο φυλακίζεται μέχρι την ενηλικίωσή του και μετά εκτελείται. Ε, οι μαστιγώσεις ή οι λιθοβολισμοί, ακόμη και σε περίπτωση βιασμού, ακόμη και σε περίπτωση συλλογικού βιασμού εφαρμόζονται. Είχαμε πρόσφατα μια τέτοια περίπτωση. Είναι μια πολύ διαφορετική κατάσταση από την παραδοσιακή και Δηλιακή που έχουμε για τις Μαλδίβες. Έχουμε λοιπόν την την ανάγκη να σκεφτούμε και να σκεφτούν και τα, τα ταξιδιωτικά πρακτορία που βάζουν πολύ διελαστικές ετικέτες και μερικές φορές οι ετικέτες αναλαμβάνουν υπόψη και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δίνω το λόγο σε έναν άλλον συντάκτη, στον κύριο Τάνοκ, για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, το 2006 ο Μοχάμετ Νασίτ, ε, εξελέχθη ως πρόεδρος μετά από 35 χρόνια δικτατορίας του κυρίου Γκαγιόμου Νασίτ, λοιπόν, προώθησε την ε, δημοκρατία, τον λαϊκισμό και προσπάθησε να εφαρμόσει το πρόγραμμα αυτό και να δώσει απάντηση σε μακροπρόθεσμα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κράτος αυτό λόγω της θέρμανσης του πλανήτη και της ανόδου του στάθμης του νερού. Σήμερα η κόρη του Γκαουγιόμι είναι η Πρωθυπουργό και ο ετεροφαλής του, αδερφός του είναι πρόεδρος και η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε συλλήψεις των ίδιων των μελών της κυβέρνησης και οι αντιπρόεδροι λοιπόν έχουν, και ο αντιπρόεδρος επίσης έχει επίσης ε, ε, συλληφθεί. Και επίσης ε, με την καταπίεση των ε, μέσων ενημέρωσης φαίνεται ότι προωθεί μία αυτοκρατία. Το σημερινό λοιπόν ψήφισμα καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να αναλογιστούν την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων κατά μελών της κυβέρνησης και των οικονομικών του συμβούλων. Οτιδήποτε άλλο δεν θα καταλήξει στην απελευθέρωση του πρώην Προέδρου Μοχάμετ Νασίδ και να επιφέρει τις αλλαγές που χρειάζεται απελπισμένα αυτή η χώρα. Ευχαριστούμε. Τώρα ένας άλλος σύντουκαν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Επίτροπε, η κατάσταση στις Μαλδίβες είναι ανησυχητική σε τρία επίπεδα. Καταρχάς, ε, επιδεινώνεται η δημοκρατία στη χώρα. Κατά δεύτερον, δεν υπάρχει αμεροληψία στους κρατικούς θεσμούς. Και τρίτον, έχουμε την ε, πολιτική υπόθεση του πρώην Προέδρου Μοχάμετ η καταπάτηση θεμελιδών ελευθεριών όπως είναι το δικαίωμα ελευθερίας έκφραση, συνάθρησης και ελευθερίας του τύπου είναι ανησυχητικά φαινόμενα και επίσης ανησυχούμε για το δικαστικό σώμα και την πολιτική διάσταση που έχει. Η διεξαγωγή της δίκης του πρώην Προέδρου Νασίδη αποτελεί απόδειξη αυτού σε μία για μια διαδικασία η οποία είναι ατελής. Και αυτό, γι' αυτό λοιπόν υπάρχει συμφωνία από όλο το πολιτικό φάσμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ζητούνται στοχευμένες ε, κυρώσεις κατά μελών της κυβέρνησης και υποστηρικτών στις Μαλδίβες. Ευχαριστώ. Η κυρία Βερζά, έχετε το λόγο ως συντάκτρια. Ευχαριστώ. Το 2008 έγιναν οι πρώτες ελεύθερες εκλογές στις Μαλβίδες. Δεν διήρκεσαν πολύ γιατί το 2012 ο κύριος Νασίτ ε, ανετράπη με πραξικόπημα. Έκτοτε οι Μαλδίβες βρίσκονται σε άθλια κατάσταση από πλευράς ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κύριος Νασίτ θα έπρεπε να μεταφερθεί στο εξωτερικό. Είναι άρρωστος. 1.200 ε, είναι οι πολιτικοί κρατούμενοι. Δυστυχώς το μορατόριο για τη θανατική ποινή ακυρώθηκε και ε, στα πλαίσια κατάπτωσης της ελευθερίας οι Μαλδίβες ε, αντιμετωπίζουν μια κατάσταση όπου αποστέλλονται πολύ στο Ιράκ σε σχέση με τον πληθυσμό. Οι Μαλδίβες εξαρτώνται από τον ευρωπαϊκό τουρισμό κυρίως και η κυβέρνηση πέρασε ένα νόμο ο οποίος απαγορεύει τον αποκλεισμό. Επίσης Υπάρχει και η ανύψωση των υδάτων που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα μέσα στα πλαίσια των κλιματικών αλλαγών. Η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει και έχει τον τρόπο της. Ευχαριστούμε την κυρία Βέρσια. Ο κύριος Παντσέρη, επίσης συντάκτης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ανησυχούμε ιδιαίτερα για την επιδίνωση της δημοκρατίας της Μαλδίβες. Επειδή υπάρχει μεγάλη καταπίεση και καταστολή των ε, μέσων μαζικής ενημέρωσης θα θέλαμε να τηρήσουν οι Μαλδίβες την απόφαση των Ηνωμένων Εθνών έτσι ώστε να απελευθερώσει τον πρώην πρόεδρο Νασίντ. Επίσης ε, θα πρέπει να υπάρχουν δίκες, δίκες με βάση τις διεθνείς αρχές περί δίκαιης δίκης και αμερόληπτης δίκης. Θα πρέπει επίσης να μην καταφέρονται οι αρχές κατά των διαδηλωτών και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κατάσταση της δικαιοσύνης και της δικαιοδοσίας στις Μαλδίβες. Θα πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στη χώρα αυτή διεθνώς. Και τώρα Ακούμε τους εκπρόσωπους των πολιτικών ομάδων από το ΕΛΚ, ο κύριος Πρέντα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν είναι η πρώτη φορά φέτος που συζητάμε την κατάσταση στις Μαλδίβες. Αυτό έγινε και προγενέστερα, όπως θα θυμόσαστε, διότι έχει επιδεινωθεί η κατάσταση στις Μαλδίβες. Στο Νασίδ, ε, στο, στις Μαλδίβες ο πρόεδρος ε, φυλακίστηκε και επειδή ακριβώς η κατάσταση υγείας του είναι πολύ κακή, θα έπρεπε να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό και όχι να παραμένει φυλακισμένος. Δυστυχώς, όπως ε, ε πρότεινε και ο κύριος θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ε, μεμονωμένες ποινές για αυτούς που πραγματικά είναι υπέτη για την απαράδεκτη κατάσταση αντιμετώπισης της αντιπολίτευσης για τα βασανιστήρια και για τον φυλακισμό των ε, ε, υπερμάχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο κύριος Χάουιτ για ένα λεπτό. Η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Μαλδίβες ε, σίγουρα δεν είναι ιδηλιακή. Ε, εκφοβισμός των ε, πολιτικών αντιπάλων, επανεφορά της ανατικής ποινής, εξαφανισμός δημοσιογράφων όπως του Αχμέτ Ριλβάν δείχνει ότι η δημοκρατία ε, υποχωρεί. Έχουμε όχι μόνο κίνδυνο των πολιτικών αντιπάλων. Με βάση διπλωμάτε, οι Μαλδίβες θέλουν περισσότερου ξένου μαχητέ κατά κεφαλή στο Ιράκ και τη Συρία από οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Πάνω από 200 τζιχαντιστέ από ένα πληθυσμό 300 και χιλιάδων φαίνεται ότι πολεμούν στο Συρία και το Ιράκ. Μας προβληματίζει η κατάσταση αυτή, η επαναφορά του Ισλαμικού νόμου, η επαναφορά σωματικών ποινών όπως το μαστίγωμα δείχνουν ε, ριζοσπαστικοποίηση και η επαναχώρηση της δημοκρατίας. Μάλιστα στο ψήφισμα του 2015 ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Υπηρετή Εξωτερικής Δράσης και τα κράτη-μέλη να εκδώσουν ταξιδιωτικέ προειδοποιήσεις προς τους τουρίστες σε σχέση με την επαναχώρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να επιβάλλουν κυρώσει σε περίπτωση που επιδεινωθούν τα θέματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φαίνεται ότι ο πρώην πρόεδρος Νασίπ βρίσκεται στον προθάλαμο της ε, εκτέλεσης. Είναι επιτέλους ε, καιρός να λάβουμε δράση για να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα αυτή. Ευχαριστώ. Mi segnalano dalle cabine della traduzione di non eh, correre troppo. Μου τονίζουν οι διερμηνείς ότι δεν πρέπει να μιλάτε πολύ γρήγορα, διαφορετικά δεν μπορούν να σας παρακολουθήσουν. Ναρτ από τους φιλελεύθερους για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα πρέπει να ε, κουράζεται ο Επίτροπος να ακούει τις ίδιες εκφράσεις όταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες οι πολιτικές ομάδες συμφωνούμε και δεν υπάρχει απόκληση. Σημαίνει ότι η κατάσταση είναι εκρηκτική. Θα ήθελα να σας πω ότι εδώ υπάρχει κατάφορη παραβίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό το ανέφεραν και οι προλαλήσαντες. Εάν δεν περάσουμε από το λόγο στην πράξη, δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να προβαίνουμε σε μία στήρα ρητορική. Γι' αυτό θα πρέπει να μην μπορούν να προσέρχονται στην Ευρώπη συγκεκριμένοι πολίτες, να παγώσουν τα περιουσιακά του στοιχεία και αυτό αφορά και την τουριστική κίνηση έναντι των Μαλδίβων. Διαφορετικά θα είμαστε υποκριτές και θα λέμε το σωστό αλλά δεν θα το πράττουμε. Η κυρία Ριβαζή έχει το λόγο για τους πράσινους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπα και οι προλήσατε συνάδελφοι, όταν βλέπουμε την εικόνα που έχουν οι Ευρωπαίοι για τις Μαλδίβες, λέμε αυτός είναι ένας παράδεισος, ένα νησί παράδεισος, ιδηλιακός. Ε, ε, αυτές είναι οι εικόνες που δίνει το Club Med ή άλλα ταξιδιωτικά πρακτορία. Για τον τοπικό πληθυσμό όμω είναι μια πραγματική κόλαση η κατάσταση στις Μαλδίβες. Πολιτικοί αντίπαλοι όπως ο πρώην πρόεδρος ε, ε, βρίσκονται στις φυλακές γιατί κατηγορούν ε, την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί ουσιαστικά το Ισλάμ όπως τη συμφέρει. επανέφεραν την θανατική ποινή. Ακόμη και 7 χρόνια παιδιά μπορούν να καταδικαστούν σε θάνατο και να μείνουν στη φυλακή μέχρι την ενηλικίωσή τους πριν εκτελεστούν. Ε, επίσης είχαμε κατάσταση εκτάτου ανάγκης ε, από την πρώην που κηρύχθηκε από την τρέχουσα κυβέρνηση. Τι θα πρέπει να κάνουμε, να πούμε στα ταξιδιωτικά πρακτορία ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προτείνουν αυτό τον τουριστικό προορισμό στους τουρίστες. Αλλά θα πρέπει και οι τουρίστες να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν θα πρέπει να πηγαίνουν στις Μαλδίβες. Μόνο ε, οι τουρίστες έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν, ε, έχουν τη δυνατότητα μάλλον να ασκήσουν πίεση, στερώντας τη χώρα αυτή από τα τουριστικά τη έσοδα. Και αν θέλουμε να εμποδίσουμε το καθεστώς θα πρέπει να επιβάλλουμε κυρώσεις οι τουρίστες να μην πηγαίνουν, αλλά και επειδή η Ευρώπη είναι ο δεύτερος εμπορικός εταίρος των Μαλδίβων, να βρούμε τρόπους να εξαναγκάσουμε την εξουσία, της ε, αρμόδιας αρχές, να επανέλθουν στο δρόμο, να δεσμεύσουμε τα περιουσιακά ε, στοιχεία των μελών της κυβέρνησης, ε, να εκδώσουμε ταξιδιωτικές οδηγίες και προειδοποίησεις. Είμαστε και εμείς, κύριε Πρόεδρε, συνυπεύθυνοι για την κατάσταση της Μαλδίβες. Κυρία Ριβαζή, υπάρχει μια ερώτηση με μπλε κάρτα, τη δέχεστε? Ο κύριος Τσαρνέτσκι. Θα Ε, συγχαρητήρια για την ομιλία σας. σας. Συμφωνώ μαζί σας. Έχω όμως μία ερώτηση. Γιατί με προβληματίζει και με ταλανίζει όχι μόνο για τις Μαλδίβες, αλλά και για άλλες περιπτώσεις. Δεν θα πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς να χρησιμοποιήσουμε και το μποϊκοτάρισμα και το τουριστικό μποϊκοτάρισμα αλλά να ασκήσουμε και πίεση, οικονομική πίεση ε, στις Μαλδίβες. Νομίζω ότι ε, η οικονομική πίεση θα ήταν η μόνη αποτελεσματική πίεση ε, που μπορούμε να ασκήσουμε και να έχει αποτέλεσμα στην κυβέρνηση των Μαλδίβων. Κυρία Ριβαζή. Συμφωνώ απόλυτα κύριε Τσαρνέτς και αυτό ακριβώς είπα και εγώ ότι είναι πολύ συνυπεύθυνοι. Καταρχήν ο κάθε ένας από εμά αν εμείς ως τουρίστες πηγαίνουμε στις Μαλδίβες γνωρίζοντας την κόλαση που βιώνει ο τοπικός πληθυσμός, αυτό μας καθιστά συνυπεύθυνου. Και τα ταξιδιωτικά πρακτορία να μην προτείνουν αυτό το τουριστικό προορισμό, γιατί έτσι ενισχύεται η παρούσα κυβέρνηση. Επίσης, αν έχουμε εμπορικές συμφωνίες με τη χώρα αυτή, να ασκούμε πιέσει μέσω των εμπορικών συμφωνιών πώς θα προχωρήσει η κατάσταση αν δεν κάνουμε τίποτα. Αν δεν κάνουμε τίποτα, αν μένουμε τα χέρια σταυρωμένα, είμαστε συνυπεύθυνοι και συνένοχοι. Όλοι πρέπει να διαδραματίσουμε το ρόλο μας. Ένα λεπτό κύριε Καστάλτο για το EFTD. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλούμε για τις Μαλδίβες κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για μια χώρα η οποία ε, ακόμα είναι παράδεισος για τον τουρισμό αλλά όμως υπάρχει πρόβλημα και δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και για τους πολιτικούς και, και για τον κόσμο. Τώρα η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει το δρόμο του αυταρχισμού και επίσης ε, έχει διαφθείρει την, τη δικαστική εξουσία και επίσης υπάρχει και Ισλαμικό κίνημα και βλέπουμε να ανεμίζουν στην πρωτεύουσα οι σημαίες ε, του Ισλαμικού κράτους. Και όλα αυτά ε, υπάρχει ακόμα το κύμα αυτό των ε, ανθρώπων που πηγαίνουν εκεί για διακοπές που τους στέλνουν οι πράκτορες. Επίσης έχουμε τόσα εκατομμύρια, τόσο κόσμο εκεί που είναι κάτω από το κατόφλι της φτώχειας. Τι θα γίνει, έχουμε και το πρόβλημα της θερμοκρασίας και έχουμε τον Νασίλ, ο οποίος ε, έπεσε ε, και θα πρέπει να περάσει από κάποια ή δίκη. Χρειάζονται επομένω κάποιες κυρώσεις για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο γίνεται, να υπάρξει εκεί πέρα ένα κράτος δικαίου. Οπότε θα πρέπει επίσης να σταματήσει και ο τουρισμός ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να βοηθήσουμε τους δημοκρατές ε, εκεί πέρα μας χρειάζονται. Πώς πίσιλ. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προσπαθούμε να τα βρούμε, να συγκεντρώσουμε μια συνένεση στο Κοινοβούλιο και να κάνουμε κάτι για όσα γίνονται στις Μαλδίβες. Να κάνουμε, όχι μόνο να μιλάμε. Και εγώ γι' αυτό σας τονίζω το εξής, ότι με ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτά τα θέματα, τα θέματα κράτους δικαίου. Και όσον αφορά αυτό το μέτωπο, στις Μαλδίβες τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Το ίδιο για τη δικαστική εξουσία και είδατε ότι έπεσε ο Νασίντ, ο προηγούμενος πρόεδρος, ε, εκτός άλλων γιατί τόλμησε να μιλήσει για διαφθορά. Επίσης, ο προϊστάμενος της Αγγελιας επάφθη παρανόμως. Συμφωνώ με όσο είπαν συνάδελφοι. Θα πρέπει κάτι να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να παγώσουμε τα περιουσιακά στοιχεία των αξιωματούχων από τη χώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενος. Κριστέα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ανησυχούμε πάρα πολύ διότι στις Μαλδίβες υπάρχει αυξανόμενη τάση να εγκαθιδρυθεί, να επικρατήσει ένα αυταρχικό καθεστώς που καταπιέζει την κοινωνία των πολιτών και τα ΜΜΕ. Ε, είναι λυπηρό αυτό, διότι μέχρι πριν λίγα χρόνια είχαμε ελεύθερες εκλογές. Ο πρόεδρος, ο παλιός, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλακή, κατηγορούμενος για τρομοκρατία. Και άλλοι πολιτικοί με τη σειρά τους καταδικάστηκαν χωρίς να υπάρξει καν σεβασμός των διεθνών αρχών περί δικαιοσύνης. Αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι η δικαστική διαδικασία ε, ε, επιτελείται χωρίς να επικρατεί η διαφάνεια. Πρέπει να δραστηριοποιηθούμε για να επηρεάσουμε τις Μαλδίβες και τη διεθνή κοινότητα, ούτως ώστε να επικρατήσει το κάτω δικαίωμα. Συνάδελφε Πόλτσακ, για ένα λεπτό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ναι αισθάνομαι υπερηφάνεια διότι βλέπω ότι υπάρχει ενότητα εδώ στο Κοινοβούλιο όσον αφορά το θέμα. Θα ήθελα να πω τι είπε ο πρόεδρος Νασίφ που ανετράπη το Φεβρουάριο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε τι συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, θα πρέπει να εκφράσουμε ένα σαφές μήνυμα που επίσης αφορά και τους δικούς μας, τους ευρωπαϊκούς λαούς. Ε, τι ελευθερίες έχουν ανασταλεί εκεί. Η ελευθερία να δρά κανείς ελεύθερα, να προστατεύεται η ιδιωτική ζωή, να υπάρχει το δικαίωμα της απεργίας, του, ε, της συνελεύσεως, ε, του να ταξιδεύει κανείς ελεύθερα από και προς το νησί. Όλα αυτά έχουν ανασταλεί όλες οι ελευθερίες οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνονται για αυτό το θέμα και να ξέρουν όταν επισκέφτονται τα νησιά τι συμβαίνει. Και θα ήθελα πράγματι τελικά να ανασταλούν οι συμφωνίες εμπορικές. Και κύριε Μπόλτσακ, έχετε μια ερώτηση για σας, δεχόσαστε. Μπονάνο, ο κύριος Μπονάνο. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Και εγώ την ίδια άποψη έχω. Η Ευρώπη όμως βλέποντας τον κόσμο. Μιλάει για ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να τα προσέχουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα συμφωνούσε να, να εγκρίνουμε την θανατική ποινή που υπάρχει στην Κίνα ή στη Σαουδική Αραβία ή να, να πάμε εναντίον τους. Μήπως θα πρέπει η Ευρώπη να μην μιλάει μόνο, αλλά να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Ή κάποιες πολιτείες, να στραφούμε εναντίον κάποιων από τις... Το, κάποιων πολιτιών την ΗΠΑ που εφαρμόζουν ε, καταδίκη. Νομίζω ότι είναι κάπως εκτός θέματος, λέει ο Πρόεδρος. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Πολτσακ να απαντήσει, ο οποίος λέει ευχαριστώ Πρόεδρε για τις ερωτήσεις. Α, χτες μίλησα για τις σχέσεις με την Κίνα. Σέβομαι την καθολική αξία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το εξήγησα. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να παραιτηθεί από το δικαίωμα να σχολιάζει με τα θέματα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ ανησυχώ και για την Κίνα και για τη Σαουδική Αραβία και για τις άλλες χώρες. Δεν θα πρέπει να σιωπάει η Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλο που είναι μεγάλη εμπορική μας εταίρια αυτές οι χώρες. Έχουμε δικαίωμα να κάνουμε την άποψή μας. Λοιπόν, πάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ορίστε κύριε Μαριά κύριε πρόεδρε οι μαλβίδες ο επίγειος τουριστικός παράδεισος προς τέρψη των ευρωπαίων και αμερικανών παραθεριστών είναι στην πραγματικότητα κόλαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. ο πρόεδρος της χώρας είχε κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης η οποία έχει αρθεί λόγω των διπλωματικών πιέσεων. το νεαρό δημοκρατικό καθεστώς στις μαλβίδες το οποίο εγκαθιδρύθηκε το δύο χιλιάδες οκτώ παραμένει εξαιρετικά ασταθές και εύθραυστο ενώ ταυτόχρονα η απειλή των τζιχαντιστών στη χώρα είναι υπαρκτή. η κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με τη διοργάνωση αντικυβερνητικών διαδηλώσεων λόγω της φυλάκισης του πρώην προέδρου της χώρας. τα ευρωπαϊκά κράτη δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουν στα εσωτερικά των τρίτων κρατών. ταυτόχρονα όμως πρέπει να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα και πολιτικά και συνδικαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα των πολιτών στις μαλδίβες οι ευρωπαίοι πολίτες οφείλουν να γνωρίζουν ότι οι ιδηλιακές παραλίες στις μαλδίβες είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου ενώ η αθέατη πλευρά του περιλαμβάνει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων φτώχεια κοινωνική εξαθλίωση και επιβολή του ισλαμικού κράτους όπου εφαρμόζεται η σαρία. ευχαριστώ η πολιτική ανάμειξη ε, στη δικαιοσύνη ε, των Μαλδιβών υπονομεύει την αξιοπιστία τους και ε, βλέπουμε να υπάρχει εκφοβισμός των αντιφρονούντων. Αυτό συνεισφέρει στην αστάθεια και στην ανασφάλεια. Η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν υποστεί σοβαρή διάβρωση με κίνδυνο να επιδεινωθούν έτσι περαιτέρω. ΜΚΟ και ε, άλλοι ακτιβιστές υφίστανται εκφοβισμό και ανησυχώ πολύ για την κατάσταση. Αυξάνεται ο αυταρχισμός, η χρήση βίας κατά ειρηνικών διατηρητών. Ε, οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν κατ' καθήκον να προστατεύουν ειρηνικούς διαδηλωτές από βίες συμμορίες. Θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά την κατάσταση και να βοηθήσουμε στη σταθερότητα την ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου με πλήρη σοβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φαντζουλικά. Ο κύριος Τελιανίδης, ο κύριος Επίτροπος έχει το λόγο. Έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Uh, Εδώ σας ομιλώ για λογαριασμό του συναδέλφου του Αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν μπόρεσε να παραστεί. Σήμερα συζητούμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Μαλδίβες. Σας ε, υπενθυμίζω ότι υπάρχει αυτή συμμαχία στα πλαίσια του COP21. Πρόκειται για τις νησιωτικές αυτές χώρες και βλέπουμε ότι μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο το κράτος αυτό στα πλαίσια της διεθνούς πολιτικής και την τελευταία φορά που συζητήσαμε για ανθρώπινα δικαιώματα στις Μαλδίβες εδώ στο Κοινοβούλιο συνέβη τούτο τον Απρίλιο. Πέρασαν από τότε 8 μήνες και η κυβέρνηση της χώρας όλο ένα και περισσότερο ακολουθεί κάποιες ε, πολιτικές που την απομονώνουν από τη διεθνή κοινότητα. Γίνεται τώρα πισωγύρισμα σε σχέση με κάποια βήματα προόδου σε ελευθερίες και δημοκρατικά δικαιώματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί κάτοικοι της χώρας που έχουν δώσει την ζωή τους σε αυτή την υπόθεση. Ε, αντιπολίτευση, ε, ελευθερία του λόγου, όλα αυτά διώκονται, οπότε υπάρχει πραγματικός ε, κίνδυνος ριζοσπαστικοποίησης της χώρας. Επίση έχουμε διώξεις και φυλακίσεις στελεχών της αντιπολίτευσης. Αυτό υπονομεύει την αξιοπιστία της κυβέρνησης και δεν είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη, οπότε αναδύονται σοβαρές αμφιβολίες για το αν υπάρχει κράτος δικαίου στη χώρα. Οπότε και ανησυχεί όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την χειραγώγηση της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση αλλά ε, όσον αφορά την εφαρμογή του συντάγματος και των νόμων. Επίσης από το βράδυ ως το πρωί η κυβέρνηση για να εξυπηρετεί φροντά της αλλάζει το Σύνταγμα. Θα πρέπει επομένως κάτι να γίνει, θα πρέπει αυτές οι αμφιβολίες να διασκεδαστούν, αυτές οι σκιές, θα πρέπει να υπάρξει κράτος δικαίου, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ούτως ώστε να υπάρξει εμπιστοσύνη προς το σύστημα και θα πρέπει να υπάρχει δίκαιη μεταχείριση όλων των κατοίκων της χώρας. Τώρα, κάποια θετικά. Ε, ισχύει το moratorium ε, de facto για την θανατική ποινή. Οπότε και εμείς ενθαρρύνουμε τις αρχές να συνεχίσουν αυτήν την πορεία. ιδίω σε περιπτώσεις που αφορούν ε, κάποιους νέους εγκληματίες, νέους τέλο πάντων καταδίκους, οριστικά να καταργήσουν θανατική ποινή και έχει ξεκαθαριστεί ότι αν δεν κάνουν κάτι τέτοιο θα υπάρξει μεγάλο πισωγύρισμα στις θέσεις, στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό το μορατό, αυτό το πάγωμα της εκτέλεσης των θανικών ποινών κρατάει επί 60 χρόνια. Η Ευρώπη παρακολουθεί το τι γίνεται σε αυτό το μέτωπο και προβληματιζόμαστε για αυτόν τον κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης στην ε, χώρα. Επίσης, πάρα πολλοί κάτοικοι των Μαλτιβών έχουν πάει να πολεμήσουν είτε με το Ζωνικό κράτος είτε με άλλους φονταμεταλιστές στο Ιράκ και τη Συρία. Συνεργαζόμαστε πάντως με την κυβέρνηση. Θέλουμε να αναδειχθούν οι βασικές αρχές ε, δημοκρατίας, κράτους δικαίου, αλλά είναι ευθύνη της κυβέρνησης να εξασφαλίσει την ασφάλεια των εκατοντάδων χιλιάδων τουριστών που πηγαίνουν για διακοπές στο αρχιπέλαγο κάθε χρόνο. Δέχθηκε η κυβέρνηση της χώρας ευτυχώ την πρότασή μας να υπάρξει κάποιος νομικός σύμβουλος που θα πάει εκεί για να αξιολογήσει την κατάσταση της εφαρμογής ε, της ε, νομοθεσίας ε, την εφαρμογή του νέου ποινικού κώδικα και ελπίζουμε ότι έτσι πρόκειται να τονιστεί σε ποιου τομεί πρέπει να γίνουν ε, βελτιώσεις και να συνάδει προς τα διεθνή πρότυπα η νομοθεσία της χώρας. Και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό βήμα από πλευράς κυβέρνησης. Έτσι θα αποδείξει ότι έχει τη θέληση να συνεργαστεί με την διεθνή κοινότητα για αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Για δημοκρατία, δηλαδή και ανθρώπινα δικαιώματα. Ελπίζουμε αυτά να υλοποιηθούν. Ευχαριστώ λέει ο πρόεδρο. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε, κύριε Στυλιανίδη. Θα είσαστε εδώ και για την επόμενη συζήτηση. Έχουμε λάβει 7 προτάσεις ε, κειμένων.